ημερήσια διάταξη θα ψηφίσουμε το, την πρόταση ψηφίσματος για το Ιράν, υπόθεση Σιρήν Εμπαντή. Τίθεται σε ψηφοφορία ένα κείμενο το οποίο ε, αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες προτάσεις. Περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται με ευρύτατη πλειοψηφία. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ψηφίζουμε έξι προτάσεις ψηφίσματος για τη Γουινέα Υπάρχει μια κοινή πρόταση που στόχο έχει να αντικαταστήσει. Δεν υπάρχει τροπολογία. Θέτω στην ψηφοφορία το κοινή πρόταση ψηφίσμου Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σας συγχαίρω και τέλος η ημερησία προβλέπει την ψηφοφορία για την ελευθερία του τύπου στην Κένια Λοιπόν γνωρίζετε τη φράση που θέλω να πω για τα ψηφίσματα αυτά και τώρα θέτω σε